Bonjour à tous. Bienvenue aux journalistes présents. Καλημέρα σας. Καλωσορίζω τους δημοσιογράφους που έχουν προσέλθει και όσους μας βλέπουν από το διαδίκτυο για να παρουσιάσουμε το αντιφασιστικό μανιφέστο και την προσυπογραφή του από ορισμένους ευρωβουλευτές. Θα με δώσω πρώτα το λόγο στην πρόεδρο της ΔΟΕ, Γκάμπι Τσίμερ. Ευχαριστώ πολύ από πλευράς της Γκουέ και Νέα ε, Ευρωπαϊκή Αριστερά του Βορρά θέλω να σας καλωσορίσω και να διευκρινίσω ότι η ομάδα της Ευρωπαϊκής Νοτικής Αριστεράς και της Βόρειας Νοτική, Πράσινης Αριστεράς θέλει να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό αντιφασιστικό μανιφέστο με βάση μια πρωτοβουλία που υπήρξε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για την καταπολέμηση του φασισμού, το ώστε να περάσει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητα. Θεωρούμε ότι δεν είναι μεμονωμένα ελληνικό πρόβλημα, που υπάρχει βέβαια η αντιπαράθεση με την Χρυσή Αυγή και η δίωξη, η ποινική για τα ποινικά εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί από τη Χρυσή Αυγή ε, κατά πολιτών, αλλά διαπιστώνουμε αυξανόμενη τέτοια δραστηριότητα στην Ευρώπη, όλο και περισσότερο διάφορες ομάδες άκροδεξιές ε, που συχνά έχουν φασιστικό χαρακτήρα σε συγκεκριμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό είναι αναγκαίο από κοινού να δημιουργηθεί ένα ευρύ πλαίσιο αντίστασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο ούτω ώστε στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη να αντιμετωπιστεί και να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε αυτές τις απόπειρες. Συμφωνούμε ότι υπήρξε όξυνση του φαινομένου λόγω του ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο ε, επιχείρησαν να αντιμετωπίσουν την κρίση, δηλαδή να τη φορτώσουν ε, στους ε, πιο απόρους και αυτό προκάλεσε κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτή είναι η κριτική μας, γιατί και πολλές κυβερνήσεις προτιμούν να επιλέξουν εθνικιστικές πολιτικές. Θέλουν δηλαδή και είναι διατεθειμένοι να αξιοποιήσουν και να στρέψουν ε, την απόγνωση ε, κάποιων πολιτών κατά κάποιων ε, στρωμάτων, εθνικών μειονοτήτων, μεταναστών, ανθρώπων που έχουν άλλο τρόπο ζωής, άλλο τρόπο σκέψης, άλλη αντιμετώπιση. Σε διάφορα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη το διαπιστώσαμε αυτό ε, τους τελευταίους μήνες. Ε, θυμίζω την αντιπαράθεση στην Ουγγαρία και τα φαινόμενα ε, εκδηλώσεων κατά τον Ρωμά που έχουμε διαπιστώσει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και είμαστε πεπισμένοι ότι χρειάζεται ένας ευρύς συνασπισμός για να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους τρόπους άσκησης πολιτικής. Πριν δώσω το λόγο στον συνάδελφο Νίκο Χουντή, θέλω να τονίσω ότι αυτές οι απόπειρες που διαπιστώνουμε από πλευράς ακροδεξιών κύκλων και άλλων, ε, α, ε, συγγνώμη, απόπειρες που γίνονται για να συγκριθούν οι, και να εξομοιωθούν οι θέσεις κάποιων ακροδεξιών ομάδων με ενέργειες και τις απόψεις της αριστεράς, αυτές οι απόπειρε έχουν οδηγήσει σε διάφορα κράτη-μέλη τα τελευταία χρόνια και τους τελευταίους μήνες, αυτές οι απόπειρες έχουν υποτιμηθεί. Δεν έχουν αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, τις έχουμε αντιμετωπίσει βάζοντάς τις κατά μέρος, δηλαδή κάποιοι εκπρόσωποι του κράτους δεν αντιμετωπίζουν ε, τα φαινόμενα δεξιάς ε, ε, βίας και εκδηλώσεων. Υπενθυμίζω πόσο χρόνο χρειάστηκε μέχρι ε, τα όργανα της κρατικής εξουσίας ή οι κυβερνήσεις να ξυπνήσουν και να καταλάβουν ότι για παράδειγμα στη Γερμανία υπάρχουν παράνομες εθνικοσοσιαλιστικές οργανώσεις οι οποίες δεν δίστασαν ακόμη και να δολοφονήσουν πολίτες που θεωρούσαν ότι δεν είναι ε, άτομα που αξίζουν να ζουν. Δεν είναι λοιπόν φαινόμενο αποκλειστικά ελληνικό, αλλά σε σχέση με την Ελλάδα είναι ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό φαινόμενο και εξέλιξη. Και θέλουμε φυσικά να σταματήσουν αυτές οι ενέργειες. Δεν θα πρέπει να αισθάνονται ότι απειλούνται ορισμένα άτομα, ότι χρησιμοποιούνται ως παραδείγματα και ως αποδιοπομπαίοι τράγοι για να αντιμετωπίσουν κάποιοι πολίτες ε, την απόγνωσή τους. Θεωρούμε ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το δικαίωμα για αξιοπρεπή ζωή για όλους τους πολίτες της Ένωσης, όλους όσους ζουν στην Ευρώπη, ανεξάρτητα από ποια περιοχή του κόσμου και της Ευρώπης προέρχονται, αυτά όλα πρέπει να τα εγγυάται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δικαιώματα λοιπόν για όλους, ανεξάρτητα αν είναι πολίτες των κρατών της Ένωσης όχι. Θα μιλήσω ελληνικά. Σας ευχαριστώ πολύ που παρευρίσκεστε σε αυτή την συνέντευξη τύπου, σε αυτή την εκδήλωση, που σκοπός είναι να παρουσιαστεί το Ευρωπαϊκό Αντιφασιστικό Μανιφέστο και να παρουσιαστεί και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αντιφασιστών Κοινοβουλευτικών. Είναι μια πρωτοβουλία αυτό το ευρωπαϊκό αντιφασιστικό μέτωπο. Είπε αρκετά πράγματα η συντρόφισσα Εγκάμπη. Εγώ υπογραμμίζω ότι η σημερινή εκδήλωση την οργανώνουμε εδώ. Μπροστά σας βρίσκονται κοινοβουλευτικοί. Συντρόφισσα Εγκάμπη που είναι πρόεδρος της Ευρωομάδας από τη Γερμανία, πρόεδρος της Ευρωομάδας της Γκουε. Εγώ ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από την Ελλάδα. Δεξιά μου η συντρόφισσα Ιανέτ Growth, δεν ξέρω αν λέω καλά το όνομα, κοινοβουλευτικό του Ντιλίνκη από τη Γερμανία. Και αριστερά, με μια ισορροπία φίλων όπω είδατε, ο σύντροφο ο Δημήτρη ο Τσουκαλά, βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου από το ΣΥΡΙΖΑ. Επομένω, είμαστε κοινοβουλευτικοί εθνικών κοινοβουλίων και Ευρωπαίων για να πούμε σήμερα ότι αυτή η πρωτοβουλία που έχει αγκαλιάσει σε αρκετές χώρες κοινωνικούς φορείς, προσωπικότητες, κινήματα. Πρέπει να στηριχτεί και είναι δική μας υποχρέωση, γι' αυτό παίρνουμε και το λόγο σήμερα, και να την παρουσιάσουμε στο Ευρωκοινοβούλιο, πράγμα που θα κάνει ο Δημήτρης και η Ανέτ, και να πούμε ότι οι ευρωβουλευτές, αντιλαμβανόμενοι ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό, να δώσουν τη δική τους υποστήριξη και να ξεκινήσουν τις δικές τους προσπάθειες, συντονισμένα και με τις άλλες και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, η σύνθεση του πάνελ, εμείς που παίρνουμε το λόγο, θέλουμε να υπογραμμίσουμε αυτή, ότι είναι πανευρωπαϊκό το πρόβλημα, η άνοδος της ακροδεξιάς, η αναβίωση του φασισμού και του νεοναζισμού, αφορά όλη την Ευρώπη. Βεβαίως δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα είμαστε εδώ από την Ελλάδα και από τη Γερμανία. Από τη Γερμανία για τους γνωστούς λόγους διότι διατηρείται ζωντανός ο αγώνας να μην ξεχαστούν τα εγκλήματα του ναζισμού και να προχωρήσουμε σε μια Ευρώπη των δικαιωμάτων, σε μια Ευρώπη της δημοκρατίας. Από την Ελλάδα, διότι έτσι ήρθαν τα πράγματα, με αφορμή την εκρηκτική άνοδο του νεοναζιστικού μορφώματος της χρυσή αυγή, που τελευταία προχώρησε και σε εγκληματική ενέργεια, προχώρησε και σε φόνο έγινε το επίκεντρο της προσοχής ή επισημάνθηκε ότι υπάρχει κίνδυνος διαμόρφωσης τέτοιων ε, φασιστικών και νεοναζιστικών οργανώσεων, εγκληματικών οργανώσεων. Αυτό που θα ήθελα εγώ να προσθέσω, δίνοντας το λόγο στη συνέχεια στον Δημήτρη και στην Ανέτ, για να μας αναλύσουν και το κείμενο και τις ιδέες, του μανιφέστο και τον τρόπο δουλειάς των κοινοβουλευτικών, είναι πως δυστυχώς χρειάζεται σημαντική προσπάθεια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε την αναβίωση της ακροδεξιάς και του φασισμού. Και χρειάζεται σημαντική προσπάθεια διότι πρέπει να αντιμετωπιστεί εκτός από τους άλλους λόγους ως αποτέλεσμα της κρίσης. Της κρίσης που πλήττει με οξύτατο βαθμό τις χώρες του Νότου μεταξύ αυτών και την Ελλάδα, από όπου προέρχεται ο Μιλών λέω για άλλη μια φορά, αλλά πλήττει μέσα από τις γενικευμένες πολιτικές της λιτότητας και τις άλλες χώρες. Και όπως γνωρίζετε η κρίση φέρνει ανεργία, φέρνει εξαθλίωση, φέρνει απόγνωση, φέρνει φόβο, φέρνει την αναζήτηση που θα στηριχτεί ο άλλος και αυτό εκμεταλλεύονται τα νεοφασιστικά ακροδεξιά μορφώματα που σηκώνουν κεφάλι στην Ευρώπη για να πάρουν την υποστήριξή τους. Και επειδή, και τελειώνω με αυτό, ο κίνδυνος περιγράφεται από πολλούς, το θέμα όμως είναι τι κάνεις, ότι πηγαίνουμε σε ευρωεκλογέ. και αυτά τα μορφώματα δυστυχώς στην Ελλάδα έχουν αποκτήσει κοινοβουλευτική παρουσία. Αύριο ενδεχομένως να έχουν κοινοβουλευτική παρουσία και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εμείς οι ευρωβουλευτές, εμείς οι κοινοβουλευτικοί, εκτός των άλλων λόγων, δεν είναι μόνο θέμα δικό μας υπόθεση, πρέπει αυτό το πράγμα να το αποτρέψουμε. Για να το αποτρέψουμε πρέπει να συμβάλλουμε σε μια ενωτική προσπάθεια, δεν είναι θέμα ελληνικό αν έρθουν από τη Χρυσή Αυγή ή αλλού, το θέμα είναι να μην έρθουν, να μην εκπροσωπούνται, να μην εκφράζουν, να μην εκμεταλλεύονται την κρίση, αλλά το χτύπημα της κρίσης, το χτύπημα αυτών των συνεπειών, ο αμήλικτος αγώνας κατά τη αναβίωσης του νοφαστικού φαινομένου να έχει και ως αποτέλεσμα να μην έχουμε τέτοια αποτελέσματα να έχει σαν συνέπεια να μην έχουμε τέτοια αποτελέσματα και στις επικείμενες ευρωεκλογέ. Αυτά ήθελα να σας πω. Επομένως σήμερα το λόγο τον έχει και τον δίνω αφού κάνουμε αυτή τη σκηταλοδρομία στο Δημήτρη τον Τσουκαλά, βουλευτή επαναλαμβάνω του Εθνικού Κοινοβουλίου από το ΣΥΡΙΖΑ, να μας πει εν συντομία όπως αυτός νομίζει γιατί είναι από αυτούς που έκανε αυτή και αυτή την πρωτοβουλία τα βασικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Αντιφασιστικού Μανιφέστου. Αν και μπορώ να μιλήσω στα ελληνικά, θα μιλήσω στα αγγλικά. Γιατί τα έχω γράψει στα αγγλικά. Φαντάζομαι θα υπάρχει μετάφραση. Θα ήθελα να πω κάτι προκαταρκτικά μετά από τα σοβαρά που είπαν η Γκάμπη και ο Νίκος. Γιατί εδώ εκπροσωπούμαστε μόνο η Ελλάδα και η Γερμανία. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολλοί και από την Αγγλία και από την Ισπανία και από τη Σλοβενία θα συμμετάσχουν, θα συνυπογράψουν το, μνημό, το μανιφέστο, αλλά ε, υπάρχουν και εμπόδια όπως η απόσταση. Τώρα όμως που είμαστε Γερμανοί και Έλληνες εδώ, η Γερμανία είχε το παρελθόν που είχε με τους Ναζί, η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα, και αυτό ακούγεται ίσως ως παράδοξο, που πολέμησε τους Γερμανούς στην κατοχή και λοιπά, στην αντίσταση. Το παράδοξο είναι ότι σήμερα έχουμε ένα τόσο μεγάλο νεοναζιστικό κίνημα στην Ελλάδα και η εξήγηση βέβαια είναι όπως είπε και ο Νίκος και η Γκάμπη προηγουμένως ότι υπάρχει πανευρωπαϊκή άνοδος του φασισμού και του νεοναζισμού. Εγώ θα περιοριστώ τώρα σε αυτά που λέει το μανιφέστο μας και ίσως να θελήσει να προσθέσει τίποτα και η Γκάμπη, αν θέλει, ως προς το πώς θα οργανώσουμε τα πράγματα. Λοιπόν, καταρχήν, το Ευρωπαϊκό Αντιφασιστικό Μανιφέστο θέλει να ακουστεί ότι υπάρχει κίνδυνος από την άνοδο της ακροδεξιά, των ακροδεξιών και φασιστικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η απειλή αυτή είναι άμεση, αλλά δεν αφορά πλέον μόνο μια χώρα όπως την Ελλάδα, αλλά όλους μας. Ποιος θα μπορούσε να πει σήμερα, ποιος τολμούσε να πει σήμερα ότι δεν είμαστε μάρτυρες εδώ στην Ευρώπη της ανάστασης, της αναβίωσης των χειρότερων εφιαλτών που έχουμε ζήσει στο παρελθόν. Ο στόχος του δικού μας μανιφέστου είναι σαφής. Να ενωθούν οι αντιφασιστικές δυνάμεις, συνδικάτα, κοινωνικά κινήματα, πολιτικά κόμματα και πάνω απ' όλα πολίτες για να δημιουργηθεί ως το δυνατόν συντομότερα ένα ενωμένο αντιφασιστικό κίνημα. Γι' αυτό δεν θέλουμε να υποκαταστήσουμε υπάρχοντα δίκτυα ή κινήματα, ούτε να διχάσουμε, θέλουμε να ενώσουμε, γιατί είναι αλήθεια περισσότερο παρά ποτέ ότι ισχύσεν τη ενώση. Μόνο ενωμένοι πέρα από εθνικά σύνορα μπορούμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες όπως την οργάνωση του ευρωπαϊκού της ευρωπαϊκής διάσκεψης ε, καλλιτεχνών κατά του φασισμού. Αυτό το ευρωπαϊκό αντιφασιστικό κίνημα πρέπει να υποφεληθεί από τις ε, ισχυρές αντιφασιστικές από το ισχυρό αντιφασιστικό παρελθόν και κληρονομιά που έχουμε, που για μερικού έχει ήδη ξεχαστεί. Δεν είναι τυχαίο ότι το μανιφέστο μας τελειώνει με τη φράση σε αυτή την ιστορική φάση δεν πρέπει να επαναληφθεί η ιστορία. Πρέπει να πάρουμε μαθήματα από την ιστορία για να μην επαναλάβουμε τα λάθη του δεκαετίας του 20 και του 30 που οδήγησαν στη χειρότερη τραγωδία της ιστορίας, την Τρεμπλίνκα, το Auschwitz και τον Παγκόσμιο Πόλεμο με 60 εκατομμύρια νεκρούς. Αν αυτό το ευρωπαϊκό αντιφασιστικό κίνημα θέλει επιτυχώς να καταπολεμήσει τον νεοφασιστικό κίνδυνο πρέπει να οργανωθεί μακροπρόθεσμα για να απορρίψει σεκταρισμούς και για να καταπολεμήσει την ακραδεξιά σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας χωρίς εξαίρεση. Και ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό είναι να απευθυνθούμε στον απλό κόσμο, στους εργαζόμενους, στον τόπο εργασίας τους. Γιατί, διότι κανείς άλλος εκτός από τον απλό κόσμο δεν μπορεί να μεταφράσει τα αντιφασιστικά τις αντιφασιστικές ιδέες σε συγκεκριμένη δράση και γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αντιφασιστών Βουλευτών που ιδρύουμε σήμερα θα είναι το πρώτο συγκεκριμένο παράδειγμα τέτοιου είδους αντιφασιστικής δικτύωσης που προτείνουμε σε όλους τους Ευρωπαίους πολίτες που θέλουν να αντισταθούν αποτελεσματικά στις νεοφασιστικές και ακροδεξιές τάσεις. Η αντίστασή μας αυτή βέβαια θα είναι δημοκρατική και θα οργανωθεί από τις ίδιες τις δημοκρατικές μάζες. Πρέπει να ομολογήσουμε αγαπητοί φίλοι ότι θα έρθουν ακόμη δυσκολότερες μέρες και ότι Τώρα είμαστε σε έναν αγώνα δρόμου κατά της βαρβαρότητας και του φασισμού. Πρέπει να οργανωθούμε και να δράσουμε τώρα και όχι αύριο. Αύριο θα είναι πολύ αργά. Παρόλα αυτά είμαστε πεπισμένοι ότι κάνουμε το σωστό. Όπως είπε και ο Γερμανός θεολόγος Dietrich Bonhoeffer, ο μόνος αγώνας που χάνεται είναι εκείνος όπου παρετούμεθα, από τον οποίο παρετούμεθα. Ευχαριστώ πριν, δώσω το λόγο στην Ανέτ. Θέλω να σας πω ότι η κυρία Τσίμερ πρέπει να φύγει γιατί πρέπει να πάει σε μια διάσκεψη για τους Κούρδους. Ευχαριστώ Φράγκο. Μια πολύ σύντομη παρατήρηση. Όπως είπαμε και προηγουμένως, πριν πάρει το λόγο ο συνάδελφός μου από τη Γερμανική Βουλή, θέλω να πω ότι είναι σημαντικό ότι είναι κοινοβουλευτικό δίκτυο. Έχουμε πολλά ευρωπαϊκά, εθνικά, διεθνικά δίκτυα κατά του φασισμού. Αλλά μέχρι στιγμής, από πλευράς ε, κοινοβουλευτικών, ένα τέτοιο ευρωπαϊκό δίκτυο δεν υπήρχε. Μετά τις επόμενες εκλογές θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι θα έχουμε πολλούς άλλους ε, ευρωβουλευτές από νεοφασιστικά κόμματα. Εφόσον αυτή είναι η εκτίμησή μας ότι αυτό θα συμβεί, τότε γνωρίζουμε ότι θα παίξει μεγάλο ρόλο πώς εμείς ως κοινοβουλευτικοί στο Ευρωκοινοβούλιο και στα Εθνικά Κοινοβούλια θα συνεργαστούμε πολιτικά. Θα έχει μεγάλη επίδραση, παραλαμβάνω. Ξέρουμε ήδη ότι πολλοί θεωρούν και από πλευρά της διοίκησης του Ευρωκοινοβουλίου ότι θα αυξηθεί κατά πολύ η εκπροσώπηση των ακροδεξιών ομάδων και επιχειρείται να τροποποιηθούν έτσι οι κανόνες για να αποφευθεί το πρόβλημα. Δηλαδή να αποκλείονται από κάποιες διαδικασίες ή να περιοθεροποιούνται από κάποιες διαδικασίες αυτοί οι ευρωβουλευτές. Παράλληλα όμως επιχειρείται τέτοιες διαδικασίες να υπάρξουν και για αριστερούς ευρωβουλευτές. Διότι αυτό ακριβώς είναι η οργανωτική αντανάκλαση της ε, εξομοίωσης των ε, ακροδεξιών φασιστικών συχνά ομάδων με κάποιες ε, ε, ριζοσπαστικές αριστερές ομάδες. Αυτό πρέπει να το καταπολεμήσουμε με επιθετικό τρόπο, να το καταγγείλουμε, να καταστήσουμε σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει υπεύθυνη αντιμετώπιση εάν η αντιμετώπιση που υπάρχει των ε, ακροδεξιών ομάδων που είναι διατεθειμένες να κάνουν εγκληματικές ενέργειες να εξισώνεται με την αντιμετώπιση σε κοινοβουλευτικό επίπεδο και εκτός των ε, κοινοβουλίων αριστερών ιδεών. Αυτό οπωσδήποτε πρέπει να το αντιμετωπίσουμε ενωμένοι, να δημιουργήσουμε ένα τέτοιο δίκτυο, να το επεκτείνουμε, να σκεφτούμε ε, εάν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα ιδρυτικό συνέδριο για να ενισχύσουμε περαιτέρω αυτή μας την πρωτοβουλία και να καλέσουμε και άλλους βουλευτές να συμμετάσχουν ούτω ώστε το θέμα αυτό κατά την προεκλογική εκστρατεία για τις ευρωεκλογέ να προωθηθεί με αποφασιστικό τρόπο ούτω ώστε μετά τις ευρωεκλογέ, αλλά και σε άλλα κοινοβούλια μετά από άλλες εκλογές όπου μπορεί να προκύψουν λοιπόν ε, ακροδεξιοί βουλευτές, ευρωβουλευτές, να κάνουμε αυτή τη διάκριση καθαρά. Να μην επιτρέψουμε να συνεχίζεται ε, αυτή η, ε, ε, η εξομοίωση. Αυτά έπρεπε να σας πω. Με συγχωρείτε που δυστυχώ τώρα πρέπει να φύγω για τις 3 η ώρα υπάρχει μια άλλη διάσκεψη ε, στην οποία πρέπει να κάνω την ανακτήρια ομιλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πρωτοβουλία. Εύχομαι κάθε επιτυχία και Ευχαριστώ πολύ τους Έλληνες φίλους που με βάση και την ε, ε, δυσάρεστη πείρα τους αποφάσισαν να θέσουν αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Η συνάδελφα μας κυρία Γκρότ. Ευχαριστώ πολύ γιατί είμαι παρούσα. Είμαι και μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και τα τελευταία χρόνια ήμουν ε, πρόεδρος ε, της ομάδας ελληνικού, ε, Ελλήνων και Γερμανών Ευρωβουλευτών στο Γερμανικό Κοινοβούλιο. Και ελπίζω να μπορέσω να διατηρήσω και περαιτέρω αυτήν την Προεδρία. Εδώ και καιρό με απασχολεί αυτό το θέμα και αυτό που με ανησυχεί ιδιαίτερα είναι το εξής. Τα ακροδεξιά φασιστικά κόμματα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο είναι πολύ καλά δικτυωμένα. Ε, όχι όμως τόσο τα αριστερά. Και διαρωτώ με γιατί. Πριν από δύο εβδομάδες περίπου δημιουργήθηκε η Αυγή στην Ουγγαρία. Μετά λοιπόν την δραστηριοποίηση της χρυσή αυγή ε, στην Ελλάδα και με βοήθεια από την Ελλάδα δημιουργήθηκε και αυτό το ναζιστικό κόμμα στην Ουγγαρία όπου υπάρχουν δύο άλλα ακροδεξιά κόμματα. Δηλαδή συνεχίζεται και διευρύνεται αυτή η προσπάθεια. Και πρέπει να υπολογίσουμε ότι θα συνεχίσει να συμβαίνει αυτό. Ότι θα αυξηθεί η επιρροή τους και θα υπάρξει μεγάλη πολιτική ομάδα και εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο ακροδεξιά. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποτραπεί κάτι τέτοιο. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε το κόμμα Φιντές, το οποίο είναι το δεξιό κόμμα της Ουγγαρίας, που είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Δηλαδή είναι στην ίδια πολιτική ομάδα με την κυρία Μέρκελ. Φέτος λοιπόν το Φίντες, αυτό το Ουγγρικό κόμμα, ε, εκφράστηκε με ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο κατά τον Ρωμά και δεν υπήρξε καμία καταγραφή κατά αυτών των ενεργειών. Πώς είναι δυνατόν να είναι μέλος του Έλκα ένα κόμμα που έχει τέτοιες απόψεις για τους Ρωμά. Έστειλα μια επιστολή στην κυρία Μέρκελ, δεν έλαβα απάντηση. Οπότε, χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτή την ελληνική πρωτοβουλία στην οποία και εγώ πολύ σύντομα, πολύ μετά την έναρξη της αποφάσισα να συμμετάσχω. Νομίζω ότι είναι καλό να υπάρξει αυτό το δίκτυο. Θα κάνω ό,τι μπορώ, ούτως ώστε και από άλλες χώρες που είναι μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης, όχι ενδεχομένω ε, της Ένωσης, να ε, συμμετάσχουν για να ενισχυθεί την προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ Ανέτ. Έχουμε ακόμη δύο-τρία λεπτά. Αν υπάρχει καμία ερώτηση λοιπόν, τώρα ας Αν όχι... Α, ορίστε παρακαλώ. Μία ερώτηση στους ε, Έλληνες συναδέλφους. Βεβαίω είναι επικίνδυνα τα φασιστικά κόμματα, αλλά δεν είναι επικίνδυνα μόνο διότι έχουν κακές ιδέες ε, και εγκληματίε οπαδούς, αλλά γιατί λαμβάνουν και υποστήριξη από διάφορους κύκλους. Άκουσα για παράδειγμα ότι στην Ελλάδα η Χρυσή Αυγή υποστηρίζεται από ορισμένα τμήματα της ελληνικής αστυνομίας και από διάφορους πλούσιους. Ξέρω ότι υπάρχουν βέβαια προσπάθειες να απαγορευτεί η Χρυσή Αυγή. Πώς βλέπετε λοιπόν την κατάσταση. Yes, this is very good question. Πολύ καλή ερώτηση. Μπορώ να μιλήσω ελληνικά. Ναι, όχι. Θα ήθελα να μιλήσω στα ελληνικά τώρα. Ε, αυτή είναι πραγματικά μια πολύ καλή ερώτηση γιατί είναι γνωστό ότι η Χρυσή Αυγή όσον αφορά τις εθνικές εκλογές είχε πράγματι μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση σε ορισμένους κλάδους της αστυνομίας. Δεν πρέπει, και η δική μας άποψη είναι ότι δεν σημαίνει ότι σύσσωμη η αστυνομία είναι με τη Χρυσή Αυγή, αλλά υπάρχουν θύλακες, υπάρχουν κομμάτια της αστυνομίας τα οποία πράγματι κοιτάζουν προς εκείνη την πλευρά και αυτό έχει πολλές εξηγήσει. Μία εξήγηση είναι αφενός μεν γιατί και οι αστυνομικοί βρίσκονται σε τραγική οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα έχουν χτυπηθεί και αυτοί ως υπάλληλοι ε, σημαντικά και βρίσκονται σε άσχημη κατάσταση. Το δεύτερο είναι γιατί επειδή η αστυνομία χρησιμοποιείται σαν ένα κομμάτι της καταστολής απέναντι στον ελληνικό λαό για να μην αντιδρά για όλα αυτά τα οποία γίνονται, δηλαδή για την πολιτική λιτότητα που υπάρχει, ε, ο λαός αντιδρά στην αστυνομία και ως καταστολή και αυτό τους ρίχνει κατά κάποιο τρόπο στην αγκαλιά της χρυσή αυγή, οι οποίοι βγαίνουν πάντα προς τα έξω υποστηρίζοντας οτιδήποτε κάνει η αστυνομία σε σχέση με την καταστολή απέναντι στον ελληνικό λαό. Άρα εδώ υπάρχει ε, κάτι το οποίο ε, εξελίσσεται, όμως έχουμε ξεκινήσει μία πορεία και μία ενημέρωση και των αστυνομικών αλλά και ολόκληρου του λαού για να κατανοήσουν και αυτοί ότι η Χρυσή Αυγή δεν είναι τίποτε άλλο από ένα κόμμα του συστήματος. Και έρχομαι στο δεύτερο σκέλος της ερώτησης, εάν υπάρχουν ε, επιχειρηματίες, επιχειρήσεις, οι οποίοι χρηματοδοτούν τη Χρυσή Αυγή. Και βέβαια υπάρχουν επιχειρήσεις. Και βέβαια υπάρχουν επιχειρήσεις που χρηματοδοτούν τη Χρυσή Αυγή, είναι εμφανές, αλλά η Χρυσή Αυγή δεν είναι μόνο ένα πολιτικό κόμμα. Είναι ένα κόμμα της νύχτας. Είναι ένα κόμμα επιχειρηματίας από μόνο του. Ασχολείται με εκφοβισμούς καταστηματαρχών, λειτουργούν ως ε, ε, σωματοφύλακες και μπράβοι διαφόρων. Άρα δηλαδή από μόνο του είναι μια εταιρεία, μια επιχείρηση καταστολής άλλων πραγμάτων. Έτσι υπάρχουν κοινές, κοινοί δρόμοι μεταξύ επιχειρήσεων και χρυσή αυγή και αυτό φαίνεται και μέσα στο Κοινοβούλιο όταν μεγάλη δηλαδή ε, όταν έχουν έρθει να ψηφιστούν νόμοι οι οποίοι ουσιαστικά βοηθούν τις μεγάλες επιχειρήσεις ή τους Έλληνες εφοπλιστές ή τους τραπεζίτες εκεί που η Χρυσή Αυγή σκίζει τα ημάτια της ότι είναι ένα αντισυστημικό κόμμα σε αυτά τα μεγάλα νομοσχέδια που εξυπηρετούν τους τραπεζίτες και τους εφοπλιστές ψηφίζει μαζί με την κυβέρνηση, ψηφίζει υπέρ των εφοπλιστών και υπέρ των τραπεζιτών. Άρα είναι ξεκάθαρο πια και αυτό είναι δικό μας θέμα. Να το αναδείξουμε στην ελληνική κοινωνία ότι είναι ένα κόμμα συστημικό, είναι ένα κόμμα όπως είναι τα κόμματα της κυβέρνησης, ε, ως προς αυτή την κατεύθυνση και δεν μπορεί να λέει ότι είναι ενάντια στη λιτότητα και ότι είναι με το λαό. Όσο περνάει ο καιρό, όλο και περισσότεροι το καταλαβαίνουν και εδώ πέρα δίνουμε μία μάχη προς αυτή την κατεύθυνση. Δύο κουβέντες συμπληρωματικά. Πράγματι, η Χρυσή Αυγή παρακολουθούντας την εγκληματική της δράση, στο στόχαστό της είχε και έχει συνδικαλιστές εργαζόμενους, μετανάστες, ομοφιλόφιλους, Ρωμά. Αυτά είναι τα θύματα της επιθετικότητας και της εγκληματικής δραστηριότητας. Δείγμα λοιπόν ότι είναι μέρος του συστήματος, κομμάτι του συστήματος και θα έλεγε κανείς και εφεδρεία του. Και το δεύτερο σε σχέση με αυτό που ισχυριστικά τώρα είναι επειδή έχουμε έναν αντίλογο. Σου λέει η Χρυσή Αυγή εμφανίστηκε, δυνάμωσε επειδή υπάρχει κρίση και σου απαντάει κάποιος. Μα κρίση έχει και άλλες χώρες. Η Πορτογαλία, η Ισπανία και δεν έχουν ένα μαζικό φαινόμενο Χρυσής Αυγής. Ή σε άλλες χώρες που δεν έχουν καθόλου κρίση. Στην Αυστρία και στην Ορθυγία, γιατί εμφανίζονται περίπου τέτοια μορφώματα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πράγματι η ερμηνεία, το πώς εμφανίζεται και σε κάθε χώρα, έχει κοινά χαρακτηριστικά, έχει και ιδιομορφίες. Γι' αυτό ακριβώς θέλουμε να φτιαχτεί αυτό το πανευρωπαϊκό μέτωπο, ούτω ώστε να είναι αποτελεσματικό να χτυπήσει τις αιτίε που γεννούν γενικά αυτό το φαινόμενο, αλλά και σε κάθε χώρα πολύ συγκεκριμένο, γιατί τότε θα είμαστε αποτελεσματικοί. Και τελευταίο, δεν ξεχνάμε η τέχνη μας βοηθάει εδώ πολλές φορές. Την ταινία του Μπερτολούτσι, 1900, πώς γεννήθηκε ο φασισμός ή πώς το αποτύπωνε, ε, πώς ο γεωκτήμονας ή και ο καπιταλιστής ε, χρησιμοποιούσε αυτούς για να χτυπήσει τους εργαζόμενους, να χτυπήσει τους αγρότες κτλ. Αυτό ισχύει και σήμερα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε χώρες που πρέπει να περάσουν ορισμένα ζητήματα. Γι' αυτό λέμε για την κρίση. Σε βάρος των εργαζομένων, των μεταναστών, των ομοφιλόφίλων κτλ. Αυτά λοιπόν τα θέματα είναι που θέλουμε να συντονίσουμε στη δράση μας για να χτυπήσουμε τις αιτίες αυτού του φαινομένου. Και το Ευρωκοινοβούλιο, επαναλαμβάνω για μια φορά, έχει και αυτό τις δικές του ευθύνες. Και η κίνηση αυτή που κάνουμε, και με αυτό, είναι μια ενωτική κίνηση. Υπάρχουν και άλλες προσπάθειες που έχουν τον ίδιο στόχο. Δεν θέλει να κλείσει αυτή η πρωτοβουλία κανενός τη διάθεση και τη δράση. Θέλουμε να ενωθούν οι πρωτοβουλίε προκειμένου να έχει το μεγαλύτερο δυνατό αποτέλεσμα εφόσον διαπιστώνουμε το τι πρόβλημα είναι αυτό, ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τι συνέπειε θα έχει για τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και γενικότερα. Ήδη έχουμε ξεπεράσει το χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μα. Θα σταματήσουμε λοιπόν εδώ. Ευχαριστώ του διερμηνείς και όλου όσου έλαβαν όλους που έλαβαν το λόγο.